πάρει αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και το λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ο κύριος Φαρή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτρο Αρία Καλμή, Ευρωβουλευτέ, τι κρίμα που δεν είναι εδώ παρόν το Συμβούλιο για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο. 25% των εκπομπών ε, ε, του θερμοκηπίου οφείλονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι κάτι ε, το οποίο ξέρουμε πόσο πολύ καταστρέφει την ατμόσφαιρα. Έχουμε τις μεταφορές τις οδικές κλπ. Το 2012 72% ήταν ε, από τις ε, οδικές μεταφορές, 12,8% ενέργειες μεταφορές, 13,9% είχαμε από τις θαλάσσιες μεταφορές. Ανάμεσα στο 1990 και το 2007 οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όλων των ε, μεταφορών αυξήθηκαν ε, πάρα πολύ. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι συνεχίζουν να αυξάνονται. Στις θαλάσσιες μεταφορές τώρα πιο συγκεκριμένα δεν έχουμε πάρει μέχρι τώρα κανένα μέτρο μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Οι στόχοι του 2020 είχαν μια ρήτρα για τις θαλάσσιες μεταφορές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις γενικές προκλήσεις. Όμως δεν έχουμε φτάσει εκεί και δεν έχουμε ακόμα διεθνείς συμφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να μειώσουμε τις εκπομπές αυτές. 4% διοξιδίου του άνθρακα εκπομπές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε τον άνθρακα να τον βγάλουμε από την ευρωπαϊκή οικονομία. Όμω δεν έχει γίνει τίποτα για τι θαλάσσιε μεταφορέ και αν δεν κάνουμε τίποτα μέχρι το 2050 οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από θαλάσσιε μεταφορέ θα έχουν αυξηθεί κατά 50%. Νομίζω λοιπόν ότι ο κανονισμό αυτό ικανοποιεί τρει στόχου. Πρώτον, ο πρώτο στόχο. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη τα οποία πηγαίνουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Είναι μια ευκαιρία έτσι να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις των ε, διεθνή Οργανισμό για τη Θάλασσα. Έτσι μπορούμε να καθορίσουμε κοινού στόχου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλή συνεργασία με τους διεθνείς μας εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό για το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα βήματα αυτά θα οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη διεθνή συμφωνία. Δεύτερον, η νομοθεσία αυτή θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα από τα σκάφη. Θα έχουμε στοιχεία με διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει να φτιάξει μια βάση δεδομένων όπου θα αναφέρεται η κατανάλωση καυσίμων από τα σκάφη. Έτσι δεν θα υπάρχουν πια βραχμοί, φραγμοί προκειμένου να οδηγήσουμε σε τεχνικά μέτρα που θα μειώσουμε τη σειρά τους στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι πιστεύω ότι θα δαπανούμε και λιγότερα για καύσιμα. Ο τελευταίος στόχος είναι ότι η νομοθεσία αυτή θα βοηθήσει να έχουμε 10.000 νέες θέσεις απασχόλησης συνδυασμένες με τις πράσινες τεχνολογίες στη θάλασσα. Καταλαβαίνω ότι το ωφέλη είναι τεράστια. Επίσης θα έχουμε μείωση των εκπομπών και όσον αφορά το μονοξίδιο του αζότου και όσον αφορά το διοξίδιο του θείου και όσον αφορά τα μικροσωματίδια. Η μείωση των εκπομπών είναι βασική προπόθεση για οποιοδήποτε άλλο μέτρο ληφθεί για τον τομέα αυτό στο μέλλον. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ που βοήθησαν τον Κρίστοφερ Φέρνερ, την Γίτε Κιούτελαν, την Γιούλι Γκέρλινγκ, τον Μπα Έικχαουτ, τον Γιώσου Γεωρητή Μπάουντ και τον Μάρκο Αφρόντε. Όπω επίση και τον πρόεδρο βέβαια, Τζοβάνι Λαβία και τον αντιπρόεδρο Μπενετικ Γιάβορ για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί. Και θέλω επίση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερο στην κυρία Μέρη Βερόνικα Πλετέσκη και την ομάδα της, το Συμβούλιο, τον Ρομπέρτο Τιλέτσε και τον Βίλεμ Μπάρκουμ που βοήθησαν πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος, ο κύριος ε, Κανέτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Φάρια, για το επικοδημητικό του έργο όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα τα μέτρα που μας προτείνει για τη δεύτερη ανάγνωση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές που βοήθησαν στην εκπόνηση του κειμένου αυτού. Πρόκειται για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα πρέπει να υπάρχει συνοχή με το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε γκρίνει για το 2030 όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα. Και δεν μπορεί οι θαλάσσιες μεταφορές να είναι ο μόνος τομέας που δεν ρυθμίζεται. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον τομέα και να μειώσουμε με χαμηλό κόστος τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το επιπλέον κόστος για την κοινοποίηση, τη συλλογή δεδομένων κτλ. σίγουρα θα αντισταθμιστεί πολύ γρήγορα. Το βασικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βρει λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τις θαλάσσιες εκπομπές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπώς θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή και να γίνεται των συζητήσεων που γίνονται στον Διεθνή Οργανισμό για τη Θάλασσα η παρακολούθηση, η κοινοποίηση κτλ. είναι ένα μήνυμα πολιτικό που στέλνουμε προς τον υπόλοιπο κόσμο, εν ώψη μάλιστα της επόμενης συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού για τη Θάλασσα που θα λάβει η χώρα το Μάιο στο Λονδίνο. Και επίση και εν ώψη τη διάσκεψη των ΗΠΑ για τι κλιματικέ αλλαγέ που θα λάβει η χώρα στο Παρίσι το Δεκέμβριο τη επόμενη χρονιά. Το κείμενο του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικό και αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχουμε πετύχει. Υπάρχει μια ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη συλλογή των πιο σημαντικών δεδομένων για το τομέα και το λιγότερο διοικητικό άχθος από τη μια μεριά διατηρούμε τον εξορθολογισμό όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, από την άλλη μεριά όμως και σύμφωνα με τόσα συζητιούνται σε διεθνές επίπεδο παρακολουθούμε τις παραμέτρους για την αποτελεσματικότητα την ενεργειακή και βελτιώνουμε έτσι βάσει των κειμένων που προτείνουν το Σεβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θέλουμε ενεργειακή απόδοση για τον τομέα που σημαίνει μέτρα και λύσεις για τον κλάδο. Ο κανονισμός αυτός διασφαλίζει ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία με νομικό πλαίσιο για ένα μελλοντικό μέτρο που θα εφαρμόζεται παγκοσμίω, τότε μπορούμε και εμείς να προσαρμόσουμε το σύστημα παρακολούθησης. Είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Έτσι προχωράμε και σε διεθνές επίπεδο με λύσεις για τον κλάδο σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ο ο πρώτο ομιλητή εκ μέρου των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Χριστόφερ Φιέλνα, για δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Οι θαλάσσιε μεταφορέ καλύπτουν ένα ποσοστό 80% των διεθνών μεταφορών. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα. Αποτελούν μέρο τη κυκλικής οικονομία. Συμβάλλουν μόνο κατά 3% στι παγκόσμιες εκπομπέ. Φυσικά και αυτό ο τομέας πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του όσον αφορά τι εκπομπέ και πρέπει να γίνουν βήματα και προκειμένου. Ελπίζω ότι τα μέτρα που προτείνουμε θα επιταχύνουν την πρόοδο προς τη μείωση των εκπομπών. Ελπίζω να ακολουθήσουν και οι άλλες χώρες γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και πρέπει όλοι να κινούμεθα με βάση τους ίδιους κανόνες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε όμως επιπλέον ότι τα μέτρα είναι αποδοτικά από οικονομική άποψη. Δεν θέλουμε να γίνουμε λιγότερο ανταγωνιστικοί ως εκ των νέων κανόνων ούτε να αυξήσουμε τον κίνδυνο τα φορτία παγκοσμίω να μεταφέρονται πλέον με λιγότερο μεταφοράς, τρόπου μεταφορά. για παράδειγμα με φορτηγά. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι καταφέραμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο διοξείδιο του άνθρακα, το πλέον επικίνδυνο αέριο, αέριο θερμοκηπίου, Χαίρομαι επίση που εξαιρέσαμε τα μικρότερα σκάφη, 40% του στόλου που όμως ευθύνεται μόνο για το 10% του συνόλου των εκπομπών. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και τέλος βεβαίω α προσπαθούμε μαζί με όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί και οι άλλες χώρες, τρίτε χώρες, πρέπει να λάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τι αναλογεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέλνα. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριο Μετέ Γκρόσε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για να επιτύχουμε μειώσει, αλλά ε, καταρχήν για να μπορεί να υπάρχει μια σύγκριση έτσι μια γενική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα. Και πράγματι είναι μικρός ο τομέας, δηλαδή το 3% των παγκόσμιων εκπομπών ε, θερμοκηπίου του άνθρακα προέρχονται από την ναυτιλία, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυξάνεται η ναυτιλία και θα είναι πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν η δική μας η πρόταση είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός για να επιτύχουμε σε τελική ανάλυση μια διεθνή συμφωνία. Προς τα εκεί πρέπει να πάει το ταξίδι, αυτή πρέπει να είναι η διαδρομή των διεθνών διαπραγματεύσεων. Ας πούμε στον ΙΚΑΟ. Ε, έχω κάνει αυτή την εμπειρία στην, στον ΙΚΑΟ. Εκεί έχουν σκληρύνει τα μέτωπα και αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις ε, κατά πόσον στις διεθνείς μεταφορές το μόνο που μπορεί να γίνει είναι ένα offsetting. Αλλά δεν μπορούμε να προχωράμε έτσι. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν και το καλύτερο απ' όλα είναι να λυθεί το θέμα ε, σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά βέβαια θα πρέπει ε, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς αν δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία. Μα αυτό το κάνουμε και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πίτροπε θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται τώρα με τη διαπραγματεύση επίπεδο IMO, ε, τι μπορούμε να περιμένουμε και έχει άραγε η Επιτροπή Plan B δεύτερη εναλλακτική λύση αν αποτύχουμε στον IMO. Δηλαδή να μην πάθουμε αυτό που πάθαμε στις ε, εναέρες μεταφορές, να ξεκινάμε, να σταματάμε και να ξαναξεκινάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια εκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, η κυρία Κέρλινγκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Η προσέγγιση του θέματος, το οποίο έλεγε στη μέση, μέρα από τον κύριο Τόπαλς, ε, δείχνει διαφάνεια, ανοιχτό πνεύμα. Ευχαριστώ γι' αυτό. Η ΣΥΑΡ θα υπερψηφίσει γιατί χρειάζεται όντω ένα σύστημα παρακολούθησης και επαλήθευσή των εκπομπών από τι θαλασσίες μεταφορέ. Ο στόχο μας ήταν ανέκαθεν ο κανονισμός να είναι εύκολος στην εφαρμογή του, να είναι αναλογικός όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις και να αποτελεί πεδίο συνεργασία με τον IMO. Μόλι ολοκληρωθούν οι συνεννοήσει με τον IMO και περιμένω και εγώ να δω που θα καταλήξουμε, τότε θα ευθυγραμμίσουμε αμοιβαίω και τι νομοθεσίε μα. Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλύτερα σε αυτόν τον τομέα, σε σύγκριση με τι αερομεταφορέ, όπου είναι μονομερή βήματα. Και εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα βήματα τα οποία αναλαμβάνει και η ναυτιλία προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρου ε, των φιλελευθέρων για δύο λεπτά, ο κύριο Νίλ Τόρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ναυτιλία... Είναι όπως οποιοδήποτε άλλος ε, τομέας πρέπει να συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Μην ξεχνούμε όμως ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος με διεθνή χαρακτήρα. Συνεπώς έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να ισχύσουν ίσοι κανόνες για όλους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό λοιπόν την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον ΑΕΜΟ, στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Είμαι ικανοποιημένος από το περιεχόμενο της έκθεσης, διότι έχει πετύχει μια ισορροπή αντιμετώπιση χωρίς να εισάγει περί τη γραφειοκρατία. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας τις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ναυτιλία ανά τον πλανήτη. Όπως είπα, έχει μεγάλη σημασία να παίζουμε όλοι με τους ίδιους κανόνες. Το αναμενόμενο, το εκτιμούμενο κόστος αυτής της υπόθεσης είναι περίπου 7.000 ευρώ ανά σκάφος, όμως ο κάθε κανόνας έχει τόση αξία ως είναι η ποιότητα της εφαρμογής του. Ας πούμε στην Βαλτική. Πρέπει να παρακολουθήσουμε όχι μόνο εμάς, αλλά και τα ρωσικά πλοία. Δηλαδή, πώς θα ελέγχουμε τα ρωσικά πλοία στην Βαλτική, για παράδειγμα. Θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Εάν ναι, τότε όντως θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και να εφαρμόσουμε εν τέλει τους κανόνες αυτούς αποτελεσματικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε περισσότερα αντί λιγότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής από την ΚΟΕ. Ε, παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ο κύριο Χωρίστη Ευχαριστώ. Με διάφορες τροπολογίες ζητάμε να διευρυνθεί το σύστημα αυτοελέγχου. Καταλαβαίνουμε ότι λήφθη η υπόψη θέση μας στην πρόταση και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τον έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας για τις εκπομπές του του άνθρακου των ε, θαλασσιών σκαφών είναι κάτι αρκετά φιλόδοξο. Θα είναι αναγκαίο. Όμως η ανταλλαγή πληροφοριών και συλλογή δεδομένων να είναι αποτελεσματική. Γιατί ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που οφείλονται στις θαλάσσιες μεταφορές θα αυξηθούν με τεράστιους ρυθμούς. Θα ουσιαστικά αντισταθμίσουν άλλα μέτρα τα οποία παίρνουμε, με τα οποία θέλουμε να μειώσουμε την θέρμανση του πλανήτη. Ο τελικός στόχος του συστήματος αυτού είναι να συνεισφέρει στην μείωση της κατανάλωσης, ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όπως λέει και ο εισηγητής, πρόκειται για ένα πρώτο μόνο βήμα. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά τη ρύθμιση και τους στόχους. Και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις στον Διεθνή Οργανισμό για τη Θάλασσα. Τέλος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρο και αν πάρουμε δεν θα φτάνει αν δεν συνοδεύεται από γενικότερο προβληματισμό όσον αφορά την ε, κατανάλωση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα για τους πράσινους ο κ. Μπαζάικου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για το ξέρω το έργο του όσον αφορά το θέμα αυτό έλαβε το έργο του κύριου Σκυλακάκη και πολύ καλά το έκανε, οπότε τον ευχαριστώ. Ε, συμφωνούμε με το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Συζητάμε τον έλεγχο, την εποπτεία ε, προς το παρόν. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η διεθνή ναυσιπλοεία ε, δεν ρυθμίζεται όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων την αναφορά των ε, στοιχείων και τη σύγκρισή τους. Είναι πολύ καλό που με τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση κατέτος να αναφέρει τα δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται μόνο για το διοξίδιο του άνθρακα. Το πιο σημαντικό ζήτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο Επίτροπος, ο κύριος Κανιέτη είναι αυτός που πρέπει να μας το πει. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι γίνεται, αλλά όλοι επίση γνωρίζουμε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ αργά. Οπότε ρωτάω τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε προκειμένου ότι ο για τη θάλασσα όντω θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα, ότι θα μειωθούν οι εκπομπέ και αν όχι, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθούν οι εκπομπέ δοξιδίου του άνθρακα των σκαφών. Γιατί πρέπει να δράσουμε. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε ο IMO μόνο να αποφασίσει κάτι, γιατί μπορεί να είναι πολύ λίγο. Προσβλέπω στις απαντήσεις σας. Κύριε Έκχουτ, υπάρχει μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Ζούλικαρτ. Δέχεστε. Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Πολύ χαίρομαι που μπορώ να ρωτήσω τον φίλο μου τον κύριο Έκχατ κάτι για αυτό το σημαντικό θέμα. Μιλάμε για τον έλεγχο, την αναφορά των δεδομένων, την επαλήθευση. Ναι. Πρόκειται για λόγια όμως. Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσθέσει και αυτό το σημείο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εν ώψη της διάσκεψης κορυφής για το κλίμα και να συζητηθεί και αυτό στη διάσκεψη στο Παρίσι και να ρυθμιστεί. Γιατί όπως είπατε και εσείς πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Μιλάμε πολύ. Ε, ήρθε η ώρα να κάνουμε και κάτι. Απάντηση Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκέρλικ για την αποτυχία της διεθνούς αεροπλοείας, εγώ το βλέπω αλλιώ. Γιατί με δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κουνήθηκε και ο υπόλοιπο κόσμος. Μερικές φορές δηλαδή βλέπετε ότι αν κάνετε εσείς κάτι, αυτό βοηθάει να κουνηθούν και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι και εδώ το ίδιο μπορεί να γίνει. Η κυρία Ντανιέλα Γιούτο, επόμενη ομιλήτρια. Ε, συγχαρητήρια και για το μωράκι σας, να σας ζήσει. Ευχαριστώ, λέει η συνάδελφος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εμείς στηρίζουμε αυτή την πρόταση κανονισμού που επιτέλους ε, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και για την ναυτιλία. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή, μάλλον η ναυτιλία συμβάλλει κατά 4% στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από τις ναυτιλιακές αρχές, από το Τάραντο, την Αγκώνα ε, και από άλλες περιοχές σχετικά με την ε, ρήπανση που προκύπτει. Και δεν είναι μόνο το διοξιδίου του άνθρακα, είναι και ακουστική ρήπανση, η χορύπανση. Πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε για να υπάρχουν καλύτερη έλεγχη αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις ε, να υπάρχει το περίφημο cold ironing που επιτρέπει ε, να χρησιμοποιούνται κάποιες συσκευές μόνο μέσα στα λιμάνια. Στην Ιταλία υπάρχουν ε, κάποιες διατάξεις που αφορούν τη χρήση αυτών των ηλεκτρικών συσκευών στα λιμάνια. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε και να εφαρμόζουμε διατάξεις χωρίς όμως να δημιουργούμε λιμάνια πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Πολύ ωραία, εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων, η επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε έναν διάλογο με καλές προθέσεις αλλά χωρίς ουσιαστικές προτάσεις. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι για την μείωση των εκπομπών. Δυστυχώς κινούμεθα πολύ διστακτικά χωρίς αποτελέσματα στην ατμοσφαιρική ρήπανση δεν κάνετε τίποτα για να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα στη ρίζα του. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που βασίζεται στι ελεύθερε συναλλαγέ. Η πρόταση που συζητούμε είναι τόσο πολύπλοκη και έχει τόσο πολύ γραφειοκρατία που δεν είναι αποτελεσματική. Το θέμα είναι οι επιχειρήσει και άλλοι φορεί να υλοποιήσουν μια αποτελεσματική μελέτη επίση την προσοχή σας στη μελέτη που αξιοποιήσαμε. Ε, δυστυχώς δεν υπάρχει μηχανισμό, διεθνή μηχανισμό που να δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να αναλάβει δράση και να πει ένα υπερεθνικό όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα για σας από την κυρία Γκραπίνη. Ε, την τάχεστε, η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφε, είστε επικριτικοί κατά της Κομισιόν. Λέτε ότι η Κομισιόν ε, δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει και δεν ε, εξασφαλίζει λύσεις. Φυσικά. Ε, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ να επικρίνουμε την Κομισιόν, αλλά έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα. Η πρόταση. Μικρόφωνο παρακαλώ. η πρόταση βασίζεται σε διαπιστώσεις και μια συμφωνία, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κενό παρόλα αυτά. Τα κράτη-μέλη κάτι πρέπει να κάνουν και να συζητήσουν διακρατικά, διακυβερνητικά και όχι σε ένα υπερεθνικό πλαίσιο. Πολύ ωραία. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Δεν θα δεχτώ άλλε μπλε κάρτε γιατί δεν έχουμε πια χρόνο. Επόμενο ομιλητή, ο κ. Τζοβάνι Λαβία, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για τη δουλειά που έκαναν σχετικά με το θέμα αυτό. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτική σημασία για την παγκόσμια οικονομία. Πάλο από 80% των εμπορευμάτων μεταφέρονται μέσω θαλάσσης. Ε, Πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι μεταφοράς και χρήση ενέργειας ε, για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, για ένα χιλιόμετρο στη θάλασσα είναι μικρότερες από ό,τι στις οδικές μεταφορές και στις εναέριες μεταφορές το 48% ε, των ε, θαλάσσιων μεταφορών βεβαίως αποδίδεται στο διοξίδιο του άνθρακα. Σήμερα το Δεκέμβρη έχει επιτευχθεί συμφωνία μετά από τις πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις με την Ιταλική Προεδρία και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα βιωσιμότητας γιατί έχει συστήσει ένα σύστημα ελέγχου για να ελέγχονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και αυτό θα χρησιμεύσει στο να οριστούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών. Να υπάρχουν μέτρα που θα είναι προσαρμοσμένα στην αγορά. Ε, να υπάρχει ένα είδος και οικονομικής αποζημίωσης. Αυτή είναι μία λύση. Ή αν θέλετε να υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων το οποίο όμως θα εγγυάται τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σε τελική ανάλυση είναι ένα βήμα προς τα μπρος όπως και αν το δει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρίστελ Σαλντεμόζε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι θαλάσσιες μεταφορές, όπως ε, προείπαμε, είναι τομέας ο οποίος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για τον περιορισμό δηλαδή των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει όσα μπορούν και γίνονται προσπάθειες. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία εμείς για τις δικές μας ναυτιλιακές εταιρείε να επενδύσουν, οι φοπλιστές να επενδύσουν σε νέα τεχνολογία. Η πρόταση που ψηφίζουμε σήμερα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα λόγω των μέτρων παρακολούθησης και επαλήθευση για όλα τα σκάφη τα οποία θα μπαίνουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συλλέξουμε στοιχεία με βάση τα οποία θα υπολογίσουμε σήμερα και στο μέλλον σε ποιο βαθμό ο κλάδος συνεισφέρει στην ρήπανση. Και τότε θα λάβουμε μέτρα. Χαίρομαι επίσης που δεν επικεντρωθήκαμε χωρίς υπάρχει λόγος στο μέγεθος τη χωρητικότητα των σκαφών, γιατί αυτό είναι μία παράμετρος και μόνο του προβλήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ένα μόνο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να συνεχίσουμε. Εργαζόμαστε υπέρ της θέσπισης παγκοσμίων προδιαγραφών, προτύπων και προδιαγραφών, παγκοσμίω όσον αφορά τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για την συμφωνία αυτή, η οποία πιστεύω ότι είναι ένα εφικτό πρώτο βήμα για να μειωθούν οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα ε, από τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, γιατί είναι το μόνο, ο μόνος τρόπος μεταφοράς που δεν έχει αναλάβει δέσμευση ε, βάσει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των εκπομπών θερμοκοπίου. Είναι λοιπόν θετικό, λάβουμε υπόψη μας ότι το 4% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα οφείλεται στις θελάσσιες αυτές μεταφορές και ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί παγκοσμίω. Άρα υπάρχει ένας αντικειμενικός λόγος για τον οποίο πρέπει και οι θελάσσιες μεταφορές να κάνουν κάποια προσπάθεια αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία αποτελούν τη βάση για, ένα, κάθε πολιτική, κάθε σωστή πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα ε, ελέγχου, αναφοράς και επαλήθευσης ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους μας. Είναι μια win-win κατάσταση και ελπίζω όλοι να στηρίξουμε την έκθεση αυτή στην ψηφοφορία σε λίγο. κυρία για μισή λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον συνάδελφό μου κύριο Φαρία. Μου είπαν ότι ήταν καταπληκτικό στις διαπραγματεύσεις. Ο προεργαλής σας ε, είπε ότι πριν από λίγο το ανέλαβε και εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος μπορούσε να τα καταφέρει ήταν αυτός που είναι Πορτογάλος. Πάντως, να πω και το εξή. Ε, για όλους μας ε, είναι σημαντικό ότι εδώ πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, να υπάρχει σύστημα ελέγχου για την αυτιλία. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την παγκόσμια προστασία προστασία του κλίματος αλλά και για τη θάλασσα. Εγώ είμαι υπέρμαχος ε, της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής και γνωρίζω ότι θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο στο μέλλον. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να προστατεύουμε το κλίμα, να μην μιλάμε μόνο για την βιοεπικιλότητα. Θα αυξηθεί η ναυτιλία κυρίως στα μεγάλα σκάφη που προκαλούν τις εκπομπές. Αυτά θέλουμε να τα καταγράψουμε και μετά να υπάρξει αναφορά για αυτά. Ε, σωστό αυτό που είπε ο συνάδελφο Ντόρμπαλτ ότι όσον αφορά τις σημαίες στην Ευρώπη όλες θα πρέπει να συμβάλλουν, να υπάρχει και έλεγχος από την Επιτροπή. Αυτό είναι δική σας δουλειά κύριε Κανιέτε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται όλες οι σημαίες. Ε, οι πλειοκτήτες ε, θα πρέπει να αναφέρονται και είναι καλό που μπόρεσε η Άλντε να πλουστεύσει τη διαδικασία σε αντίθεση με την πρόταση Επιτροπής. Καλό που υπάρχει διαφάνεια και που αφαιρούνται ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα. Γενικά πρέπει να πω χαίρομαι πάρα πολύ που Ευρώπη προχωράμε και ε, προσπαθούμε να επηρεάσουμε το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO. Ε, στις περιοχές ΖΕΚΑ με εκπομπές ε, θείου, αν το καταφέραμε να το επιτύχουμε και, εκεί, αυτό, αυτό θα ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Πολύ ωραία. Η κυρία Κίλενεν είναι η επόμενη μιλήτρια. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ το πρωί κυρία Πρόεδρε οι διεθνείς ε, θαλάσσιες μεταφορές ε, είναι ο τρόπος μεταφορών ε, που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω της νέας οδηγίας περί εκπομπών θείου. Έχουμε λοιπόν τώρα την οδηγία ΣΕΚΑ και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανανεώνεται ο στόλο και η τεχνολογία. Όσον αφορά τώρα τη θάλασσα θα μπορούσα να σας ε, πω πάρα πολλά αλλά νομίζω ότι στην κοινοβουλευτική μας εργασία θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το χειμώνα η θάλασσα καλύπτεται από πάγο και κατόπιν του τα σκάφη μπορούν ε, να την διασχίσουν μόνο με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια και αυτό είναι πρόβλημα στις ε, μελλοντικές μας εργασίες. Ε, προφανώς και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, να μην αγνοούμε θέματα ασφάλειας. Ευχαριστούμε όλους, λέει η Πρόεδρος, που τηρούν το χρόνο που έχει προβλεφθεί για εκείνους. Επόμενη για 1,5 λεπτό, η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο στόχος μας είναι μια διεθνής συμφωνία με την οποία θα θεσπίζονται οι κανόνες για όλους. Η αρχή είναι καλή πάντως. Στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Διεθνής Επιτροπή όπου συμμετέχω ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Είναι ο μόνος τομέας που δεν καλύπτεται από συμφωνία ή κανόνες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέτρα εμπροκειμένου. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλουμε να τρώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εφοπλιστές πρέπει λοιπόν με βάση την πρόταση να υπολογίσουν το ποσό των εκπομπών για κάθε διαδρομή. Να αναφέρουν λοιπόν στοιχεία σε αιτήσια βάση, κατά το οποίο όλοι το θέλουμε τους ή άλλως. Και μετά η και κάθε δύο χρόνια θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. είναι ο στόχος, αλλά πρέπει να συμμετάσχουν προκειμένου και οι τρίτες χώρες. Διότι, για παράδειγμα, στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, στο, του πρόβλημα δηλαδή τι γίνεται με τα μεγάλα κροσγερόπλια Και αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμεί. Επόμενη, κυρία Μίρια Μιτάλε, για λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ολλανδικά έχει. Όχι. Η πρόεδρος, η πρόεδρος διακόπτη, μισό λεπτό, <laughs> είμαστε αναγκασμένοι να σας ε, ε, διακόψουμε γιατί δεν υπάρχει διερμηνία. Μήπως μπορείτε να περιμένετε λιγάκι. Μήπως μπορείτε να ξαναξεκινήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι το 2011 είχαμε τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για τις Μεταφορές που έλεγε ότι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα προς θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον 40% μέχρι το 2050 αν τις ε, συγκρίνουμε με το 2005. Στην πραγματικότητα, παρά την εισαγωγή ελάχιστων μέτρων ενεργειακής απόδοσης για νέες κατηγορίες σκαφών και παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, φαίνεται ότι εκπομπές από τα σκάφη στη θάλασσα θα αυξηθούν. Ίσως γιατί το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνει. Η αύξηση αυτή των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα των πλοίων δεν ευθυγραμμίζεται βέβαια καθόλου με τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το πρώτο θετικό βήμα είναι οι διαπραγματεύσεις με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Θάλασσα προκειμένου να μειωθούν παγκοσμίως οι εκπομπές αυτές. Έτσι θα μειωθούν γενικότερα οι εκπομπές εφόσον βέβαια ε, ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και υπάρξει κατάλληλη τεχνολογία για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Είναι κάτι θετικό σίγουρα. Όλοι οι τομείς πρέπει να συνεισφέρουν στη μείωση της ύπασης της ατμόσφαιρας. Και αν λάβουμε υπόψη μας τη διεθνή διάσταση των ε, θαλάσσιων μεταφορών, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η μείωση αυτή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συμφωνία στον IMO και καλό θα ήταν να ξέρουμε ο IMO τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποχτάνιο ε, για ένα λεπτό και εκείνος. Κύριε Επίτροπε, οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι μόνος τομέας που δεν καλύπτονται από κανόνες όσον αφορά την υποχρέωση μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης και επαλήθευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι βεβαίω σημαντική. Δεν καταλαβαίνω όμω, γιατί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τι ευθύνε τη και δεν απαιτεί τα αντίστοιχα από τους άλλους. Αλλιώς θα βρεθούμε σε δινή θέση από πλευρά ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος για τον τομέα, για τον κλάδο αυτόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίση κίνδυνο να μεταφέρουν τα πλοία του οι σε άλλε σημαίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να επιβαρύνουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία συμπεριλαμβανομένη φυσικά τη ναυτιλίας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Η επόμενη μιλητήρια, κυρία Καγιακάλα για ένα λεπτό. Είναι σημαντικό φυσικά να είμαστε πρώτοι στον αγώνα προστασία του κλίματος. Όμως, ας μην βλάψουμε τι εταιρείε μα προσπάθεια μείωσης των εκπομπών πρέπει να είναι παγκόσμια. Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Ο ανταγωνισμός δεν είναι τοπικός, αλλά διεθνής. Οι διατάξεις για το θείο, για παράδειγμα, στην Βαλτική αύξαν το κόστος των θαλασσίων μεταφορών και αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνούμε ότι οι επιχειρήσεις μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικές διεθνώς και ότι κάποια στιγμή κάποιοι, κάποιες θαλάσσιες οδοί μπορούν να εκπέσουν για να υποφεληθούν άλλοι. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν παραμένει σημαντικό μέλημα. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρο. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτο ομιλητή είναι ο κύριο Ζαν Κέλλη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Και εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόταση. Κάτι πρέπει να γίνει, επιτέλους, για τις εκπομπές ε, της ναυτιλίας. Από τον κλάδο των θαλασσιών μεταφορών. Εάν παραμείνουμε απραγή η ρήπανση θα αυξηθεί. Αν κάνουμε κάτι Λοιπόν, θα κινηθούμε προς την σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι και το μήνυμά μας. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Φυσικά, αυτά τα οποία κάνουμε, είπε και ο Επίτροπος, μάλιστα όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς σημαντική επιβάρυνση. Τα σχετικά κόστη είναι μικρά. Έτσι, κάνοντας το πρώτο βήμα, δίνουμε και το παράδειγμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και μη ευχαριστούμε ο κύριος Ρικάρντο ο Σάντος για ένα λεπτό. Ε, Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι η κύρια αιτία εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αλλαγές γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο και σίγουρα αλλάζει και σύνθεση των ωκεανών μας εξαιτία των εκπομπών αυτών. Γι' αυτό και πρέπει να μειωθούν επιγόντως, κυρίως εκείνες που οφείλονται στη θάλασσα στις θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είτε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε άλλα καύσιμα, τα οποία καταστρέφουν λιγότερο το περιβάλλον. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιούμε με ορθολογικό τρόπο, με λογικό τρόπο το καύσιμα. Στη, στα μέση του Ατλαντικού μπορούν να γίνεται να παίρνουν καύσιμα τα πλοία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο κύριος Διάκοπιτς επίσης για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που ήδη γνωρίζετε. Η Κροατία είναι χώρα με θαλάσσιες μεταφορές. Για μας θαλάσσιες μεταφορές είναι σημαντικός οικονομικός τομέας και έχουμε μεγάλα λιμάνια που είναι πολύ σημαντικά για μας ε, και είναι ναυπηγική ε, και αυτή παίζει ρόλο στην οικονομία μας. Έτσι λοιπόν όταν ε, μιλάμε για αυτόν τον κανονισμό νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και για την ρήπανση που προκαλούν. Δεν θα πρέπει να μετράμε μόνο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και άλλου είδους εκπομπές. Και είμαι ευγνώμων σε όσους συνέβαλαν στο να επιτευχθεί αυτό το συμβαστικό κείμενο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τον τομέα της εναυπηγική και άλλων ε, βιομηχανικών τομέων. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι θαλάσσιες ε, μεταφορές θα επεκταθούν κατά πολύ στο μέλλον ως εμπορευματικές μεταφορές. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτόν τον τομέα όπως επίσης και τα καύσιμα που καταναλώνονται στον τομέα αυτό. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες προτάσεις, παρήματος χάρη όσον αφορά τη χρήση φυσικού αερίου αλλά και τη χρήση νέας μορφής καυσίμων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να εισάγουμε νέα συστήματα εμπορίας φυσικού αερίου και να σκεφτούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόμακρες ε, περιοχές. Να βελτιωθούν και οι συγκοινωνίες ανάμεσα στα νησιά και από τα νησιά προς την Ήπειρο. Και αυτό τόσο όσον αφορά τις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές μεταφορές. Τελευταίος ο μιλητής στη διαδικασία Catch the Eye, ο κύριος Νίκολα Καπούτο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι οι μόνες μεταφορές ε, που ε, δεν ελέγχονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα παρότι συμβάλλουν κατά πολύ και στην ατμοσφαιρική ρήπανση και στην αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου. Εμερεβού αυτό είναι το σύστημα για να ελέγχονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Ευρώπη θα εφαρμόσει πολιτικές μείωσης ε, των εκπομπών του άνθρακα να ελέγχεται η ατμοσφαιρική ρήπανση η επεξεργασία λοιπόν μιας φιλόδοξης πολιτικής όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών σε αυτόν τον τομέα είναι ακόμα πιο σημαντική έχοντας κατά νου τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι θαλάσσιες μεταφορές κατά τα επόμενα χρόνια. Ε, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός άρα δηλαδή είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξουν πράσινες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται οι υδρογονάνθρακες ε, αλλά και άλλα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το λόγο και πάλι ο κύριος Κανιέτα και σας παρακαλώ πολύ αν είναι δυνατόν κύριε Πίτροπε να τηρήσετε τα δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το σημαντικό τους έργο. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα σημαντικό μήνυμα που συνάδει με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το πακέτο ενέργεια και κλίμα ε, με στόχο το 2030. Σίγουρα και ο θαλάσσιος τομέας πρέπει να συνεισφέρει στην μείωση των κλιματικών αλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει συνολικά λύσεις όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη θάλασσα. Σίγουρα πρέπει να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα στην διάσκεψη στο Λονδίνο το Μάιο του Διεθνούς Οργανισμού για τη θάλασσα, αλλά και στα τέλη της χρονιάς στο Παρίσι. Χρειάζεται ένα σύστημα παρακολούθησης, κοινοποίησης, σύγκριση των δεδομένων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα, αλλά αποτελεί και μια σημαντική θετική εμπειρία στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων. Όταν συζητάμε αυτά τα θέματα σε διεθνές επίπεδο, η εμπειρία μας θα βοηθήσει να εντοπίσουμε λύσεις που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Εξάλλου, και μια που τηρούμε την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο να προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου στη θάλασσα θα φροντίσουμε σε διεθνές επίπεδο να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα και εφόσον υπάρξει διεθνώς θα προσαρμόσουμε και εμείς το δικό μας ε, το σύστημα. Διακόπτη η Πρόεδρος. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέρφους παρακαλώ ησυχία για να μπορούμε να ακούμε τον Επίτροπο. Μην κάνετε πηγαδάκια εδώ στο ημικύκλιο όσο μιλάει ο Επίτροπος και στη συνέχεια ο εισηγητής. Αν θέλετε συζητήσεις μεταξύ σας, εκτός ημικυκλίου παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, συνεχίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποιοι ευρωβουλευτές ρώτησαν σε ποια κατάσταση βρίσκονται διαπραγματεύσεις στον IMO. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης, κοινοποίηση και επαλήθευσης σε διεθνές επίπεδο. Προχωράνε αργά, αργά, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κοινοτική νομοθεσία που έχουμε μπροστά μας αποτελεί όθηση στην διαπραγματευτική διαδικασία. Η Προεδρία του Παναμά, εξάλλου, είναι αισιόδοξη όσον αφορά τη διαδικασία. Όμως, τώρα που μιλάμε και έτσι όπως έχουν διαπραγματεύσεις, φαίνεται δύσκολο, αν και όχι αδύνατο, να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις πριν το Παρίσι. Γιατί υπάρχουν χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, που εξακολουθούν να έχουν θέσεις που δεν διευκολύνουν τη συνολική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα. Πρόεδρος Διακόπτη, συνάδελφοι, ακούστε παρακαλώ και μην μιλάτε όσο ε, έχει το λόγο ο Επίτροπος και στη συνέχεια γιατί συγγνώμη κύριε Επίτροπε που σας διακόψα αλλά έπρεπε. Τελευταίος τώρα ο εισηγητής μας, Ιγνάσιο Φάρια, για δύο λεπτά. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Microphones, for the technician. Ε, το μικρόφωνο παρακαλώ. Okay. Okay, it seems we have a technical problem. Από ό,τι φαίνεται έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. It's fine. Can you try again, Mr. Farias? Ε, μήπως μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε, κύριε Φαρίας. Commissioners. Ε, δυστυχώς το μικρόφωνο του Επιτρόπου, μάλλον το μικρόφωνο του Επιτρόπου έχει κλείσει, ίσως μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιο άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, οι τεχνικοί έχουν την καλοσύνη να κλείσουν το μικρόφωνο στο κέντρο εδώ υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ο κύριος Φαρίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την τελική φάση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και τον Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω να ακούτε παρά το γεγονός λοιπόν ότι ε, τον ε, ομιλητή τον ε, επιβαρύνουν νέες υποχρεώσει γιατί στο μέλλον θα γίνεται για την διαβίβαση και τον έλεγχο των δεδομένων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνεται έλεγχος η ενέργεια κατανόλωνεται και το καθεξής. Αυτές οι διατάξεις ε, ε, προφανώς και θα συνεπάγονται διοικητικό άκτος και θα ήθελα να πω το εξή. Κοιτάξτε, στο μέλλον θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που ήδη υπάρχουν από τα σκάφη και με τον τρόπο αυτό αυτά θα είναι σκάφη το 55% του στόλου μιλάμε για αυτά που εκπέμπουν ε, διοξίδιο του άνθρακα και κατά τα άλλα θα παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο πλαίσιο του IMO. Ε, και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πιστεύω ότι αυτές οι διατάξεις είναι πολύ σημαντικές για τον τομέα της ε, ναυτιλίας και επίση και για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ένα σημαντικό πρωτοβήμα στο οποίο θα ακολουθήσουν και επόμενα έτσι ώστε να αφαιρέσουμε το διοξίδιο του άνθρακα από τις ε, μεταφορές και ελπίζω αυτό να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως ε, μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, δεν μπορέσαμε γενικώ να παρεμποδίσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, όμως μπορέσαμε να θέσουμε ένα γενικότερο στόχο ε, και αυτό επιτεύχθηκε με τη συνένεση των κομμάτων, επιτύχαμε το συμβιβασμό. Ελπίζω λοιπόν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας θα εισακουστεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επιτέλους ε, συμφώνησαν, επικράτησε η λογική και ελπίζω λοιπόν ότι τώρα πια ε, θα εγκριθεί η πρότασή μας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι που δείξατε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και ελπίζω να συμφωνήσετε με την πρότασή μας. Ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Φάρια. Ε, φαντάζομαι Χαρήκατε τουλάχιστον ε, να μιλήσετε εδώ από το μικρόφωνο της Επιτροπής. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Ελπίζουμε και οι τεχνικοί να ελέγξουν κάπως ε, το πρόβλημα. Έκλεισε λοιπόν η συζήτηση και ε, σε λίγα λεπτά ξεκινάει η ψηφοφορία.